πρακτικά. Και ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση Ντεχάνε και Κάλφιν σχετικά ε, με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι ονομαστική ψηφοφορία και είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισαν λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι. Ερωτώ για άλλη μια φορά. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Κατόπιν τούτου έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση. Πάμε τώρα στην έκθεση Τρασκόψκη. Υπαριθμόν ένα τροπολογία. Όλες οι τροπολογίες ψηφίζονται με ονομαστική ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν ψηφίζουμε για τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Υπαριθμών 2 αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, το 3, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 4, αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Γίτσες και πάλι γίτσες λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, γκρίνεται, αλλά φτάνει τώρα. Πάμε τώρα στην υπαριθμόν 4. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η υπαριθμόν 5. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα η παριθμόν 5 στο πρωτότυπο κείμενο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η παριθμόν 6. Αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία υπερθμών 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο της πρότασης. Ο κύριος Κάρας παρακαλώ έχει το λόγο. Πρέπει να ανακοινώσω ότι δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε καμία ψηφοφορία ε, διότι δεν λειτουργεί το, η συσκευή που έχω μπροστά μου. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε τώρα ονομαστικά, χωρίς τον κύριο Κάρας. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Και πάμε τώρα στην έκθεση Λαβία. Διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάλι έκθεση Λαβία για τον διορθωτικό προπλησμό υπαριθμών 8. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάμε τώρα στην έκθεση Πλένκοβιτς. Το λόγο με βάση το άρθρο 138 έχει ο εισηγητής. Ο εισηγητής παρακαλώ. Δεδομένου ότι δεν έχει προβλεφθεί συζήτηση για την έκθεση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΛΚ που μου ανέθεσε την έκθεση αυτή. Είναι η πρώτη μου έκθεση. Είναι και η πρώτη έκθεση ενός Κροάτη Ευρωβουλευτή. Πρόκειται ε, για την κατάσταση στη Βαλένσια και έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συνάδελφε, χαίρομαι πάρα πολύ που ευχαριστείτε το ΕΛΚΑ, αλλά εξ όσων γνωρίζω, οι συγητέ ορίζονται από το Κοινοβούλιο και όχι από τι μεμονωμένε πολιτικέ ομάδε. Αλλά παρόλα αυτά, ευχαριστούμε πολύ που εσεί ευχαριστήσατε. Ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον συνάδελφο Πλένκοβιτς. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Πακ σχετικά με το πρόγραμμα Έρασμος για όλους. Καταρχήν λοιπόν θα ψηφίζουμε για την υπαριθμόν 1 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν καταπίπτουν όλες οι άλλες ε, τροπολογίες και Ψηφίζουμε για την τροποποιημένη ε, πρόταση επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και η νομοθετική πρόταση, η μονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Πακ. Πάμε στην επόμενη έκθεση, η κυρία Κώστα, έκθεση Δημιουργική Ευρώπη. Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Ψηφίζουμε για τον μπλοκ υπερθμών 1, σύνολο Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει τον μπλοκ υπερθμών 2. Ψηφίζουμε για την τροποποιημένη πρόταση επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομοθετική πρόταση με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Η ψηφοφορία έκλεισε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον, στην εισηγήτρια, στην εισηγήτρια, στην κυρία Κώστα. Πάμε τώρα στην επόμενη έκθεση, Τάκουλα πριν από την ψηφοφορία ο εισηγητής ε, θέλει το λόγο επιδιαδικαστικού. Παρακαλώ κύριε Τάκουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο εισηγητής ε, του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020 θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω ξανά τις πεπιθήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο κανονισμός αυτός βρίσκει την τέλεια λύση για τη σύνδεση με τον πολιτισμό και την ιστορία όπως προβλέπονται στο άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν αυτό αποτελεί νομική βάση. Έπρεπε να έχει εφαρμοστεί σωστή νομική βάση για την νομοθετική διαδικασία για αυτό το φάκελο. Ο μόνο λόγο για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκατέλειψε τη θέση του για την νομική βάση και δέχτηκε τη διαδικασία συνένεσης ε, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν βάσει του άρθρου 352 ήταν ότι επιθυμούσε να αποφύγει το πολιτικό διαδικαστικό αδιέξοδο και να καθυστερήσει τη θέση του προγράμματος. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν ήθελε να ξαναπροκύψει μια τέτοια κατάσταση Προτείνω αυτή η δήλωση να προσαρτηθεί στο νομοθετικό ψήφισμα. Okay, vielen Dank. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάκουλα. Ψηφίζουμε τώρα για την τροποποιημένη πρόταση στην υπαριθμόν φορά στη νομική βάση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έτσι λοιπόν οι τροπολογίες 2-106 καταπίπτουν και περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, έκθεση της κυρίας ε, των κυριών Βαλεάν Ρικέα ή άλλα Ζέντα. Καταρχήν ψηφίζουμε για τη συμβαστική πρόταση την 135 ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιπε ε, τροπολογίες καταπίπτουν και πάμε στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις εκθέσεις, στην έκθεση των κυρίων Κουμουτσάκου και Ερτούγκ. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κουμουτσάκο, έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από δυόμιση χρόνια σκληρής δουλειάς, ψηφίζουμε σήμερα και με την ψήφα μας κάνουμε ένα ποιοτικό, ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα προόδου για τις μεταφορές στην Ευρώπη ανταγωνιστικότητα ανάπτυξη απασχόληση είναι ο τριπλός στόχος που επιτυγχάνουμε με τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. ένας στόχος ζωτικός για την ευρωπαϊκή οικονομία για τους ευρωπαϊκούς λαούς ειδικότερα για τις χώρες συνοχής και εκείνες από τις χώρες μέλη που όπως η χώρα μου υφίστανται μια βαθιά ύφεση και μεγάλη ανεργία. θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για τη σημερινή επιτυχία. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουμουτσάκο και περνάμε στο μπλοκ υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν όλες οι υπόλοιπες ε, τροπολογίες καταπίπτουν και περνάμε στην τροποποιημένη πρόταση επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην έκθεση Δεκάστρο. Μπλοκ υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου, το μπλοκ υπαρτιμών 2 καταπίπτει και υπέρ τη τροποποιημένη πρότασης επιτροπή, κατά παρακαλώ, Αποχέ. εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον κύριο Ντεκάστρο. Και πάμε τώρα στην έκθεση Scholz. Πρόκειται για τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον κύριο Σόλτ. Και περνάμε στην έκθεση του συναδέλφου Γκρούτε. Μία και μόνο ψηφοφορία έχουμε. Όσοι παρακαλώ συμφωνούν με την έκθεση Γκρούτε, να σηκώσουν το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Πάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Ρέμεκ. Συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ΙΤΕΡ. Ψηφίζουμε λοιπόν για τι ε, τροπολογίε τη ε, κυρία Επιτροπής 1, 7, 9, 16, 18, 24 υπέρ παρακαλώ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ, αν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τοπολογία υπαριθμών 8. Έκλεισε η ψηφοφορία. Οριακή η πλειοψηφία. Εγκρίνεται πάντως. Τροπολογία υπαριθμών 35 και η 31 κατόπιν του καταπίπτουν και πάμε στην 32 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθμών 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου η τροπολογία υπερθμών 33 καταπίπτει. Περνάμε στην 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 30 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται και πάμε στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Υπάρχει μία τροπολογία, 27 ε, αναθεωρημένη, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στο νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή τον κύριο Ρέμεκ. Πάμε τώρα στην έκθεση Σκίνερ. Ψηφίζουμε για τις ε, τροπολογίες της κύριας επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ. Κοιτάξτε, ξαναρωτάω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 90 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 91 δέλτα, ντε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογίες 24-32 της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ή εγκρίνονται. 92 D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 33 έως 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 93 έως 96 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε υπέρ, ε, το έχω πει, έκλεισε η ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος, ψηφίσατε όλοι, απορρίπτονται και συγγνώμη ζητώ. Η 101 αναθεωρημένη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κυρίε και κύριοι, θέλω να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται το δεξί χέρι κουράζεται όλο και περισσότερο. Και αυτό μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν μπορώ να δω ότι ψηφίζετε. Πάμε τώρα στην 97. Υπέρ. Κατά. Ωραία λοιπόν. Αποχές. Απορρίπτεται ή 98 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 68 και η 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 δέλτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 89 ε, δέλτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, μισό λεπτό λέει Πρόεδρος. Πάμε στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα και αυτό με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Κράμερ και ψηφίζουμε για τις τροπολογίες επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η 6 σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ για το πρώτο, υπέρ κατά, αποχές ε, εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα, ε, υπέρ κατά, αποχές ε, πρέπει να έχουμε ηλεκτρονική επανήθευση. ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ξανά. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 33, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η 18 υπέρ μισό λεπτό ε, κατέπεσε η 18 εφόσον εγκρίθηκε η 33 κατέπεσε η 18 περνάμε στην 29 ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται η 30 επίσης με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 31. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 32, επίσημα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η έκθεση του κυρίου ε, Κράμερ έγινε δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Και τώρα πάμε στην έκθεση Τσίτσεστερ. Και ψηφίζουμε για τις τροπολογίες της κύριας Επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ. Ξαναρωτάω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται ή εγκρίνονται η 39 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 40 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 41 επίσης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 25 υπέρ μισό λεπτό Εφόσον έγινε δεκτή 42, κατέπεσε 25, πάμε στην 38 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται και νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση.